Buenos días a todas Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους. Damos comienzo la, la reunión eh, Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση με τις ανακοινώσεις της Προεδρίας, της Προέδρου καλύτερα. Ελπίζουμε, ή μάλλον δεν μπορέσαμε να τελειώσουμε τους συντονιστές λόγω χρόνου. Υπάρχουν όμως κάποιες ε, προτάσεις προς τις ομάδες σε σχέση με το πρόγραμμα εργασίας για το 2016 και για τις εκθέσεις τις οποίες ε, θα προωθήσουμε τον επόμενο χρόνο. θα υπάρξει ενημέρωση των πολιτικών ομάδων από τους συντονιστές και θα συνεχίσουμε με το θέμα αυτό γιατί όπως σας είπα δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε σήμερα το πρωί την ε, συνεδρίαση. Το επόμενο θέμα είναι η πρόταση χρονοδιαγράμματος των συνεδριάσεων για το 2016. Έχετε τις πληροφορίες αυτές στην διάθεσή σας. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, πολλά θέματα εδώ να συζητήσουμε, αλλά <clears throat> νομίζω ότι μπορείτε να εγκρίνετε εφόσον το επιθυμείτε το χρονοδιάγραμμα το οποίο σας προτείνουμε. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια αμφιβολία ή κάποια διαφωνία. Και περνάμε στις ψηφοφορίες αμέσως. Πρώτη έκθεση προς ψηφοφορία είναι ο γενικός προϋπολογισμός. Enmienda número 1, votos a favor. Ποιοι είναι υπέρ το 1, κατά, αποχές δεκτή η 1, τροπολογία 2 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές θα υπάρξει ηλεκτρονικός έλεγχος λέει η Πρόεδρος του δεύτερου τμήματος της τροπολογίας υπαρίθμου 2. Ψηφίζεται. Sí, se rechaza Λοιπόν, το δεύτερο τμήμα ε, δεν έγινε δεκτό. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 3 και εδώ κατά διαίρεση ψήφος. Πρώτη υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Αν θέλετε να υπάρξει έλεγχος στο δεύτερο τμήμα της τροπολογίας υπαρίθμου 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. ...21 ψήφοι υπέρ, 6 ψήφοι κατά. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν Βλέπω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τέσσερα Πέρα στις ψηφοφορίες. Απερίφθη. Η 6 τώρα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Α, συγγνώμη, λάθος, έκανα 5, η τροπολογία 5, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. Τροπολογία 6 λοιπόν, πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτό. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα της 6. Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη το δεύτερο τμήμα. Η 7. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή οι 8 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Η εννέα υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. δέκα υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη και τώρα η τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά πέρα της ψηφοφορίας 23 ψήφοι υπέρ, 5 ψήφοι κατά. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία της επόμενης έκθεσης Ουρτασούν για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις προτεραιότητες για το 2015. Θα ξεκινήσουμε με την τροπολογία 19. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές, απερίφθη. Α, έλεγχος. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 19. Τέλος. Απερίφθη. Λοιπόν, η δική μου ψήφος, ε, δεν έχω την κάρτα μου, αλλά είναι κατά. Λοιπόν, η 20, ποιοι είναι υπέρ. Η 20, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι η ίδια ψηφοφορία με την προηγούμενη. Τέλος. 13 υπέρ, 14 κατά και μία αποχή απερίφθη η 20. 21 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 22 άρχεται η ψηφοφορία Πέρασης ψηφοφορίας Συγγνώμη. <clears throat> Υπάρχει άλλη μια συνάδελφος χωρίς κάρτα. Απερίφθη εν πάση περιπτώσει. 23 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε τώρα στην 30 σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ κατά, αποχές, δεκτό. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος για το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Δεκτή. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 34 και 35 ταυτόσημες. Ψηφίζουμε μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 34 και 35. Ψηφίζεται. Τέλος. <clears throat> Δεκτή. 36 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 36 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτή. Περνάμε λοιπόν τώρα στην 40. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος Είναι λίγο θολά τα πράγματα, δεν μπορώ να διακρίνω, οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Δεν ξέρω αν κάποια ομάδα άλλαξε άποψη, μάλλον ε, δεν έπεσα τόσο έξω. Λοιπόν, 41 υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Περνάμε στην 47 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος στη 47. Πέραστη ψηφοφορίας. Απερίφθη. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 48 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 52 σε 2 τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απερίφθη. Περνάμε στην 53 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 57 σε 2 τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για τη συμβιβαστική 2 ψηφίζεται απερίφθη η συμβιβαστική απερίφθη Τρία υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τρία άρχεται η ψηφοφορία τέλος Τέσσερα υπέρ α συγγνώμη έγινε δεκτή η τρία καταπίπτει η τέσσερα. Περνάμε στην 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την 11 ψηφίζεται τέλος της ψηφοφορίας απερίφθη 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος στο δεύτερο τμήμα της 13 ψηφίζεται Τέλος. Απερίφθη. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δε, απερίφθη α, ηλεκτρονικός έλεγχος πάλι για την 18 άρχεται η ψηφοφορία πέρα της ψηφοφορίας απερίφθη έτσι κι αλλιώς απερίφθη λοιπόν. Αξεχάσαμε την τροπολογία 15. Παρακαλώ πρέπει να ψηφίσουμε τη 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. 21 υπέρ 6 κατά. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία των τελικών τροπολογιών για τον ρόλο των Ηνωμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη. Παρακαλώ να ψηφίσουμε en bloc όλες μαζί τις τροπολογίες, όχι. Λοιπόν, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 3, υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και τώρα θα ψηφίσουμε την προφορική ερώτηση για τους στόχους του προηγούμενου προγράμματος Δάφνη. Ισότιμα δικαιώματα κτλ. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τέλος ε, με τις ψήφους.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 Eh, λοιπόν, κανονικά θα ξεκινήσουμε στις 11. Πρέπει να είναι εδώ η συγγήτρια, γύρω από την οποία και την έκθεσή της θα γίνει το hearing. Θα διακόψουμε λοιπόν μέχρι τις 11. Χρόνος να πιείτε ένα καφέ. καπό μας

AUTHORWAVE

Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ξεκινάμε την ακρόαση για την ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο. Και ο Όπως γνωρίζετε, στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου πήραμε την απόφαση να οργανώσουμε κάποιες ακροάσεις σχετικές με τις εκθέσεις πρωτοβουλίας τις οποίες έχει ψηφίσει η Επιτροπή μας. Στην παρούσα φάση ασχολούμεθα με το θέμα αυτό η έκθεση της κυρίας Ρέτνεκ, έκθεση πρωτοβουλίας, θα μας ε, κάνει λοιπόν μια εισαγωγή η κυρία Ρέντκε. Ευχαριστώ εδώ και τους τρεις ομιλητές, τις τρεις ομιλήτριες μάλλον, οι οποίες θα συνεισφέρουν στη συζήτησή μας. Να σας θυμίσω ότι έχουν συγκεκριμένο χρόνο οι ομιλίες σας, όχι πάνω από 10 λεπτά, για να μπορέσει να ακολουθήσει μια κάποια συζήτηση με, τις, ε, με τους ευρωβουλευτές άνδρες και γυναίκες. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Σραμ που ασχολείται με τα θέματα του ίντερνετ. Έχετε το λόγο κυρία Σραμ για 10 λεπτά. Hello. Καλημέρα σας. Hello, yeah. yes. So, hi. Um, I'm... Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Τζούλια Σχάμ. Είμαι πολιτική επιστήμων και συγγραφέα και εργάζομαι για το Ίδρυμα Μαντέου Αντώνιο που είναι μια πρωτοβουλία για την κοινωνία των πολιτών και την δημοκρατική κουλτούρα. Θα σας μιλήσω για την ε, ε, ρητορική μίσους και το μισογενισμό στο διαδίκτυο. Το 2015 γίνεται λεώνα και σαφέστερο το τι σημαίνει η ψηφιακή αλλαγή για την κοινωνία και για την επικοινωνία. Δηλαδή, ο πολιτικός διάλογος έχει γίνει πιο δημοκρατικός. Όμως ο πολιτικός διάλογος ήταν ε, αποκλειστικό προνόμιο των ε, παραδοσιακών ε, μέσων ενημέρωσης. Τώρα όμως με την ε, ψηφιακή εποχή έχει δοθεί βήμα σε περιθωριοποιημένες μέχρι πρώτη ομάδες. Για παράδειγμα υπάρχει το hashtag στο Twitter κραυγή στα γερμανικά όπου γυναίκες μπορούν να μιλήσουν για περιστατικά σεξουαλικής παραενόχλησης και δυστυχώς αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν όλο ένα και συχνότερα. Η ρητορική μίσους είναι ένα φαινόμενο που έχει αυξηθεί και έχει γίνει πραγματικό πρόβλημα στα κοινωνικά μέσα και ε, παρεμποδίζει το δημοκρατικό διάλογο. Η πολυμορφία κινδυνεύει από αυτή τη ρητορική μίσους. Όμως, ακριβώς λόγω της εκδημοκράτησης ε, του διαδικτύου και του πλουραλισμού στο διαδίκτυο ακούγονται πολλές ε, φωνές που μέχρι προτενώς δεν μπορούσαν να ακουστούν. Ο σεξισμός ε, έχει γίνει πλέον θέμα συζήτηση στην ψηφιακή εποχή. Πολλοί είναι οι λόγοι. Καταρχάς οι γυναίκες χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα πολύ περισσότερο από ε, πριν και συνεχίζει να αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν πλατφόρμες όπως το Instagram όπου το 80% των χρηστών είναι γυναίκες. Εκεί λοιπόν οι γυναίκες μοιράζονται σκέψεις, ανησυχίες για διάφορα γυναικεία θέματα, σεξουαλική παρενόχληση ή ε, πιο πρόσφατα συζητιέται το θέμα της μητρότητας και το ότι πολλές γυναίκες έχουν μετανιώσει που έκαναν παιδιά. Είναι κάποια θέματα λοιπόν τα οποία ε, συζητώνται στα κοινωνικά μέσα, τα οποία μέχρι πρώτη θεωρούνταν ε, ταμπού. και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ο σεξισμός και ο ρατσισμός λοιπόν έχουν γίνει θέματα συζήτησης. Για παράδειγμα η ράπερ Μινάς αναφέρεται σε αυτά στη δουλειά της και δημόσια. Αυτή λοιπόν η οργάνωση των γυναικών δεν είναι αρεστή σε πολλούς άντρες. Αυτή η οργάνωση που γίνεται στο διαδίκτυο έχει αντίδραση. Οι γυναίκες δεν ε, μπορούν πλέον να σοπάσουν και δεν τους ενδιαφέρουν οι αντιδράσεις των ανδρών. Και εδώ αρχίζει η ρητορική μίσους. Έχουν αναδυθεί διάφορες ε, ομάδες ε, που διακρίνονται από μισογυνισμό, από σεξισμό και στοχεύουν γυναίκες οι οποίες έχουν γνωρίσει επιτυχία. Ένα παράδειγμα είναι το λεγόμενο Gamergate. Είναι αυτό το σκάνδαλο το οποίο έχει και παραπομπές στο Watergate, όπου λοιπόν, τι έγινε, μία νέα γυναίκα ε, είναι σχεδιάστρια βιντεοπαιχνιδιών, έχει φτιάξει ένα παιχνίδι για την ε, κατάθλιψη και έχει λάβει καλές κριτικές. Ε, εμφανίστηκε όμως ένας άντρας, ο πρώην της έτσι όπως ισχυρίζεται, ο οποίος προσπαθεί να την εκδικηθεί και την διαβάλλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις το θέμα αυτό τον τελευταίο χρόνο και αυτό έχει οδηγήσει σε μία τρομακτική αύξηση περιστατικών σεξισμού στο διαδίκτυο. Έχω συλλέξει κάποια παραδείγματα για να σας δώσω το μέγεθος του μισογενισμού που επικρατεί στο, στην ψηφιακή εποχή και στα ψηφιακά μέσα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες ε, γυναίκες, δύο πολύ γνωστές γυναίκες ε, σχεδιάστριες παιχνιδιών, οι οποίες έχουν ε, λάβει απειλές ακόμα και για τη ζωή τους στο διαδίκτυο και στην Wikipedia μάλιστα. Όπως βλέπετε στη διαφάνεια, μία γυναίκα, η Μπραϊάννα Γου, έπρεπε να φύγει από το σπίτι της γιατί τη συνέβη αυτό που ονομάζουμε στο διαδίκτυο doxing, δηλαδή η αποκάλυψη της πραγματικής της ταυτότητας χωρίς τη θέλησή της. Η γυναίκα αυτή ασκούσε κριτική πάνω στον σεξισμό που επικρατεί στην ε, βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών και αυτό φυσικά είχε αντιδράσει. Κάποιοι άρχισαν να τη γράφουν ότι ξέρουμε ποια είσαι, που μένει, δημοσίευσαν τα στοιχεία τη, την ξεμπρόστιασαν δηλαδή, έκαναν απειλέ για τη ζωή τη, για τη ζωή των δικών τη. Και η τελευταία, το τελευταίο στιγμιότυπο οθόνη, ε, βλέπετε εδώ. Λέει ότι θα αρχίσω να, ε, να παίζω Grand Theft Auto μόνο και μόνο για να αρχίσω να βαράω γυναίκες. Βλέπετε λοιπόν το μέγεθος του σεξισμού που υπάρχει στο διαδίκτυο. Δεν θα σας δείξω τα χειρότερα, αλλά είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι συντονισμένες επιθέσεις κατά των γυναικών, οι οποίες αυξάνονται στο διαδίκτυο και είναι μισογυνισμός άνευ προηγουμένου. Πολλές γυναίκες έχουν βρεθεί σε αυτή τη θέση και χρησιμοποιούν τα κοινωνικά μέσα έτσι ώστε να χειροφετηθούν, να ενισχύσουν τη θέση τους και να αντιδράσουν σε αυτή τη ρητορική μίσους, ε, του μισογυνισμού. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει κοινωνικός διάλογος όχι μόνο στα κοινωνικά μέσα αλλά και αλλού. Στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης αυτό το θέμα έχει αποσιοποιηθεί. Τώρα όμως το διαδίκτυο μας δίνει τη δυνατότητα να το συζητήσουμε. Η ρητορική μίσους είναι κάτι που ε, πλήττει περισσότερο τις γυναίκες, περισσότερο τους ε, έγχρωμους από ότι τους λευκούς, περισσότερο τους ομοφιλόφιλους από ότι τους ετεροφιλόφιλους. Ε, ε, η ρητορική μίσους είναι ενδεικτική της ισορροπίας των δυνάμεων στην κοινωνία μας. Χρειάζεται να αναλυφθεί δράση, διότι κάθε επίθεση δεν πρέπει να παραμείνει ε, χωρίς αντιμετώπιση. Επίσης υπάρχουν και άλλα φαινόμενα, υπάρχει η παρενόχληση στο διαδίκτυο, το cyberbullying και επίσης αυτή η παρενόχληση λαμβάνει χώρα εντός συγκεκριμένου πλαισίου, όπου οι άνθρωποι αυτοί παρενοχλούνται ε, από τους ε, συνανθρώπους τους. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο εκφοβισμός, ο οποίος μπορεί να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις και μάλιστα οδηγεί σε αυτό που λέμε στα γερμανικά shitstorm, δηλαδή χαμός παίρνει τεράστιε διαστάσεις, φεύγει εκτός ελέγχου και μάλιστα οι κοινωνιολόγοι ε, λένε πως ε, όλα αυτά μπορούν να προκαλέσουν μετατραυματικές ε, διαταραχέ, όπως μια ληστεία ή ένας βιασμός. Αυτέ λοιπόν είναι οι ακραίες εκφάνσεις της ρητορικής μίσου στο διαδίκτυο. Επίσης υπάρχουν απειλές για βιασμό, απειλές για τη ζωή κάποιου, η αποκάλυψη ιδιωτικών ε, στοιχείων και πληροφοριών όπως ε, τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, ε, διεύθυνση, εκδικητική πορνογραφία μετά. Όλα αυτά συνδέονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Τι, τι είναι η εκδικητική πορνογραφία λοιπόν. Είναι η δημοσίευση γυμνών φωτογραφιών γυναικών από τους πρώην συντρόφους τους στο διαδίκτυο έτσι ώστε να ντροπιάσουν την γυναίκα. Πολλές φορές αυτό έχει ως αποτέλεσμα να λάβουν απειλές για τη ζωή τους ή ε, να παρενοχλούνται συστηματικά. Αυτές λοιπόν οι επιθέσεις είναι συντονισμένες και είναι πραγματικά αποτελεσματικές, ε, οδηγούν τις ε, γυναίκες σε αποκλεισμό. Πολλές γυναίκες έχουν εγκαταλείψει τον ακτιβισμό εξαιτίας αυτών ακριβώς ε, των μισογενιστικών πράξεων. Και πραγματικά ποιος θα περίμενε πως το διαδίκτυο θα είχε τόσο μεγάλη δύναμη. Είναι λοιπόν ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο χρήζει αντιμετώπισης. Πώς όμως, καταρχάς πρέπει να πούμε πως η λογοκρισία και ο περισσότερος έλεγχος δεν θα λύσει το πρόβλημα, θα κάνει μάλιστα το αντίθετο. Υπάρχει δυσανάλογη, δυσανάλογος βαθμός διακρίσεων απέναντι στις γυναίκες. Πολλοί θεωρούν πως είναι ε, ανώφελο να κάνουμε κάτι, διότι κανείς δεν μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες, κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Τώρα, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη ρητορική μίσους. Χρειάζονται ιδιωτικές πρωτοβουλίες, ε, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, χρειάζεται αντίδραση της κοινωνίας των πολιτών. Η ρητορική μίσους πρέπει να βρει αντίδραση, πρέπει να αντιμετωπιστεί ανοιχτά και όχι να καταστέλλεται. Επίσης υπάρχουν διάφορες, ε, διάφοροι άλλοι τρόποι αντιμετώπισης, η διαγραφή και ο αποκλεισμός των χρηστών που... Ε, γράφουν με τέτοιο τρόπο από τα κοινωνικά μέσα για παράδειγμα. Η καταπολέμηση της ρητορικής μίσους στα κοινωνικά μέσα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο διότι είναι διάσπαρτη και κατακαιρματισμένη. Δεν μπορούμε λοιπόν να ε, την αντιμετωπίσουμε χωρίς πολύ καλό συντονισμό. Η άγνοια πρέπει να καταπολεμηθεί έτσι ώστε να καταπολεμηθεί και ο σεξισμός. Πρέπει αυτό όπως σας είπα να ε, γίνει στα πλαίσια μιας συντονισμένης αντίδρασης και όχι μεμονωμένων ενεργειών, διότι μόνο έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Τα σχολεία, το εκπαιδευτικό σύστημα επίσης μπορούν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο αυτό, διότι ε, διαφορετικά κινδυνεύουν να ενταθούν αυτές οι διαφορές. Τέλος, τουλάχιστον ε, το διαδικτυακό πλαίσιο χρειάζεται χρηματοδότηση πρωτοβουλειών οι οποίες θα ε, ασχοληθούν με την ε, ενημέρωση σχετικά με τα φαινόμενα μισογενισμού και σεξιστικής βίας στο διαδίκτυο. Χρειάζεται λοιπόν ενημέρωση και όχι άμεση καταπολέμηση, διότι όπως σας είπα δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Χρειάζεται εκπαίδευση από νεαρή ηλικία, χρειάζεται κατάρτιση των ε, αστυνομικών αρχών έτσι ώστε να ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα διακρίσεων και ρητορικής μίσου στο διαδίκτυο διότι πολλές φορές οι αστυνομικές αρχές δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν και συχνά πολλές φορές η μόνη απάντηση που έχουν στα θύματα είναι εντάξει μην χρησιμοποιείτε το ίντερνετ τότε. Φυσικά πρέπει να στηρίξουμε την, ε, τις προσπάθειες σε όλη την Ευρώπη κατά πολέμησης του σεξισμού κυρίως στο διαδίκτυο διότι εκεί είναι το πεδίο μάχης. Εκεί θα κρυθεί λοιπόν ο πόλεμος. Αυτά λοιπόν από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και θα ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον τα επόμενα σχόλια και τις παρεμβάσεις. Ευχαριστώ κύριε Σραμ. Το λόγο τώρα θα το δώσω στην κυρία Μπερζέ. Uh, first I would like θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε και το θερμό όρισμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερους την Κωνσταντς Λεγκρίπ που με προσκάλεσε στη σημερινή ακρόαση. Θα συνεχίσω στα γαλλικά. Euh, Συνεχίζω λοιπόν στα γαλλικά. Το πρώτο που μου φαίνεται πολύ μεγάλη σημασία σε, όταν μιλάμε για την ισότητα των δύο φύλων είναι ότι ο βασικός αγώνας που πρέπει να κάνουμε είναι να κατακτήσουμε έδαφος. Περί αυτού πρόκειται όταν μιλάμε για την ισότητα των δύο φύλων. Κερδίζουν όλο ένα και περισσότερο έδαφος κατακτώντας το χώρο που τους αναλογεί στο δημόσιο βίο. Διότι ε, δυστυχώς εξακολουθούν να επικρατούν εκεί οι άντρες. Οι γυναίκες παραδοσιακά στριμώχτηκαν, εγκλωβίστηκαν ένα λεπτάκι να βάζω και τις διαφάνειες ε, ταυτόχρονα γιατί προσπάθησα να ε, φέρω και λίγο το χιούμορ στην παρουσίασή μας ε, στη σημερινή ακρόαση. Έλεγα λοιπόν ότι ε, στην, στον ιδιωτικό ή ακόμη και στον οικιακό χώρο είχαν εκλοβιστεί για πολύ καιρό οι γυναίκες ε, και στο δημόσιο χώρο ήταν μόνο περαστικές. ενώ οι άντρες μπορούσαν να σταθμεύουν και πέρα. Το βλέπουμε. Είδατε και τις εικόνες νωρίτερα στο μετρό είχε γίνει ολόκληρη ε, εκστρατεία ενημέρωσης για να κατακτήσουν και πάλι το χώρο που τους αναλογεί χωρίς ακόμη και στα μέσα μαζικής ε, μεταφοράς. Ε, το βλέπουμε και στις γειτονιές μας. Οι άντρες επικρατούν σε αυτό το χώρο και δεν θεωρείται θεμητή κατά κάποιο τρόπο η παρουσία των γυναικών εκεί. Πολλοί θέλουν να εκλείψει η γυναίκα ή να την κρύβουμε. Ή ακόμη ε, προτιμότερο να εξαφανιστεί και να μην εμφανίζεται καθόλου σε δημόσιους χώρους. Υπάρχει και ένας ε, νέος αγώνας λοιπόν για την επανάκτηση αυτού του δημοσίου χώρου που γίνεται στο διαδίκτυο, στο web ακόμη ευρύτερα. Υπάρχει λοιπόν ένας ψηφιακός χώρος έκφρασης ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ε, στα κοινωνικά δίκτυα, στα φόρες, στα blog. Πέρα από την έκφραση όμως διαμορφώνεται και η κοινή γνώμη. Ε, και πολύ εύκολα μία γνώμη γίνεται πλειοψηφική τη σήμερα. Ας πάρουμε και το παράδειγμα τη ΣΥΣΚΟ. Δημιουργείται και ένας νέος οικονομικός χώρος στο ιστορικό του ψηφιακού χώρου και, έχει, και λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη για την καινοτομία αλλά και κομιστής ενός νέου τρόπου διάρθρωσης ε, των ε, κοινωνικών ε, σχέσεων αλλά και των σχέσεων στον χώρο εργασίας. Σε αυτό το δημόσιο χώρο έχουμε διαφορετικές ταυτότητες, έχουμε την ψηφιακή διάσταση αλλά και την οικονομική διάσταση. Παρόλα αυτά βλέπουμε ε, ότι υπάρχουν ε, στερεότυπα και πρέπει να διαπιστώσουμε εάν καταργούνται παλιές παραδόσεις, αν γίνονται νέες προσπάθειες για να υπάρξει μια κοινή ε, κατάληψη αυτού του ψηφιακού χώρου σε αντίθεση με το παρελθόν. Εσείς, ε, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπατε, ασχοληθήκατε με αυτό το πρώτο ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να επικεντρωθώ ε, στις ε, ευκαιρίες, στις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται σε αυτό το ψηφιακό χώρο. Δεν ξέρω αν είδατε αυτό το εξώφυλλο του Newsweek που σχολιάστηκε πάρα πολύ ε, για τις γυναίκες τη Silicon Valley. Το Newsweek ήθελε να αρθρογραφήσει λοιπόν για αυτές τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο Silicon Valley Είναι λίγο σεξιστικό το εξώφυλλο, αλλά έκανε το γύρο του κόσμου. Βλέπουμε λοιπόν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τα στερεότυπα και οι προκαταλήψει, συγγνώμη, ε, εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητες, όμω υπάρχει μια νέα γλώσσα. Ο ψηφιακό ε, κώδικα που πρέπει όλοι να μάθουν, υπάρχει άνηση μεταχείριση, το βλέπουμε ως προ τι αμοιβέ ε, και κυρίω το βλέπουμε σε αυτόν τον οικονομικό χώρο στο, στον επαγγελματικό προσανατολισμό των γυναικών και ε, στενεύει ακόμη το περιθώριο για τις γυναίκες να ακολουθήσουν ε, επιστημονικούς κλάδους ε, στη Γαλλία. Παραδείγματος χάρη μόνο 10% ασχολούνται με την ανάπτυξη λογισμικών και ασχολούνται με τις νέες τεχνολογίες, τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Οι ευκαιρίες όμως, οι νέες ευκαιρίες υπάρχουν και είναι στο γενετικό κώδικα του web. Κατάργηση των συνόρων πρώτα απ' όλα. Το ψηφιακό χώρος εξορισμού δεν οργανώνεται πλέον κάθετα αλλά οριζόντια. Άρα επιτρέπει παρίσφρηση ε, με μαζικό τρόπο και ε, με ταχύς ρυθμούς των γυναικών σε αυτό το χώρο ε, ενώ παραδοσιακά αποκλείονταν από οποιοδήποτε χώρο εξουσίας. Στο Κοινοβούλιο επίσης ε, κάνετε ε, συχνά συζητήσεις για την ουδετερότητα του web. Ε, πάλι στον γενετικό κώδικα του web υπάρχει γενής αυτή η ιδιότητα της ουδετερότητας και μπορούμε εμείς να την αξιοποιήσουμε. Πώς μπορούμε λοιπόν να δράξουμε αυτές τις ευκαιρίες και να μετατρέψουμε αυτό το ε, αυτά τα γενετικά χαρακτηριστικά του web σε νέες ευκαιρίες ε, για τις γυναίκες. Πώς θα αγωνιστούμε σε αυτό το νέο χώρο για να καταπολεμήσουμε τα στερεότυπα. Θα βασιστούμε στην αρχή ότι εξακολουθούν να υπάρχουν Άρα πρέπει και εμείς να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να τα καταπολεμήσουμε αυτά τα στερεότυπα ε, εις ε, του, των γυναικών. Επίσης, στον ψηφιακό χώρο υπάρχει ε, ένα διπλό ε, μειονέκτημα για τις γυναίκες ε, υπάρχει το σύνδρομο της απάτης ε, και μιλάμε για τις νέες τεχνολογίες και για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, αυτολογοκρίνονται οι γυναίκες και θεωρούν ότι δεν έχουν κάποια θέση σε αυτό το χώρο όπου πνευματικά και οικονομικά επικρατούν οι γυναίκες ε, και έχουν το σύνδρομο της κατωτερότητας, αν θέλετε, Υπάρχουν πρωτοβουλίες όπως η Duchesse France παραδείγματος χάρη. Είναι ε, όμιλοι που καθημερινά αγωνίζονται ούτω ώστε ε, στην, στις νέες τεχνολογίες και στους επιστημονικούς κλάδους να μπορέσουν επίσης να ε, εισχωρήσουν σε αυτό το χώρο και οι γυναίκες ε, ούτως ώστε με αποτελεσματικότητα να καταπολεμήσουμε αυτό το σύνδρομο διότι αυτή τη στιγμή το εντοπίσουμε το σύνδρομο και το δεχτούμε μπορούμε να το ε, γιατρέψουμε. Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα στη Γαλλία ε, στο, το, για το βούτυρο. Σε αυτό το τομέα υπήρξαν πάρα πολλές ε, δυσκολίες ε, και δημιουργούνται νέες πρωτοβουλίες και άρα προκύπτουν και νέες οικονομικές ευκαιρίες. Αυτό που σήμερα συμβαίνει με το βούτυρο μπορούν να συμβεί και με άλλες πρωτοβουλίες για τις γυναίκες. Εγώ δεν θέλω να κάνω αυτή τη διάκριση ανάμεσα στις ευκαιρίες για τις γυναίκες και τις ευκαιρίες γενικότερα για την καταπολέμηση οποιασδήποτε διακριτική μεταχείρισης. Είναι αυτό που συμβαίνει. Αν δείτε ε, ποιοι είναι οι υποψήφοι και ποιοι είναι ε, αυτοί που από γίνονται επιχειρηματίες, ε, είναι αυτοί που μακροχρόνια είχαν αποκλειστεί από, τον, από την αγορά εργασίας. Έτσι, στον ψηφιακό χώρο με νέες ευκαιρίες μπορούμε ταχύτερα, με, με μεγαλύτερη προβολή με πιο μαζικό τρόπο να μπείτε σε αυτόν τον απαγορευμένο μέχρι τούδε κύκλο. Το είπατε κι εσείς ε, νωρίτερα, υπάρχει φυσικά ε, ε, εδώ το ζήτημα της εκπαίδευσης, κατάρτισης της παιδείας. Υπάρχει και το θέμα του ε, σχετικού ε, ψηφίσματος του ΟΗΕ για τις γυναίκες. Είναι η νέα γλώσσα που πρέπει να μαθαίνουν. Αν τους το αρνηθούμε αυτό, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του 21ου ε, αιώνα. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για την παραδοσιακή παιδεία και κατάρτιση. Η εκμάθηση του, ε, της ψηφιακής γλώσσας από πρώιμη ηλικία πρέπει, ε, είναι κάτι το απαραίτητο πλέον. Είναι μια νέα γλώσσα την οποία απλώς πρέπει να διδάξουμε στο σχολείο και δεν έχει σχέση μόνο με τον ψηφιακό χώρο. Ο στόχος είναι να ενσωματώσουμε τον νέο τρόπο προσέγγισης αυτής της γλώσσας και αυτού του κόσμου, αυτού του νέου κόσμου, μέσα από τη γλώσσα του. Ε, όταν μιλάμε για τις ε, προκλήσεις λέμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει αυτό σε μικρή ηλικία και κυρίως για τις γυναίκες. Πέραν αυτού σε όλες τις χώρες δεν πρόκειται για αναπτυγμένες είτε για αναπτυσσόμενες. Το θέμα της εκμάθησης αυτού του κώδικα και ε, το, ο αλφαβητισμός, ο ψηφιακός αλφαβητισμός είναι βασικές προϋποθέσεις εκ των νόν ουκάνευ. Δεν μπορεί να θεωρείται πλέον ως gadget, ως κάτι περί το πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως βασική προϋπόθεση προϋπόθεση για την παιδεία εν γέννη. Και επιμένοντας σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το νέο δημόσιο χώρο που δημιουργεί τις νέες ευκαιρίες διότι είναι κομιστής όπως είπαμε αυτών των νέων ευκαιριών εγγενώς έχει αυτές τις νέες ευκαιρίες Αναγάγοντας λοιπόν αυτήν την ε, μάθηση της ψηφιακής γλώσσας σε μια βασική προϋπόθεση, με ταχύτερο τρόπο, με μεγαλύτερη προβολή των αναγκών θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ισότητα των δύο φίλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βερζέ. Η τελευταία ομιλήτρια τώρα. Η κυρία Μόρου από την εταιρεία Cisco. Δεν έχω διαφανίες, θα πρέπει να με ακούσετε. Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, εξ ονόματος της ΣΥΣΚΟ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας σήμερα είναι κάτι το οποίο συνοδεύει φυσικά και έρχεται αμέσως μετά τη μεγαλύτερη μεταναστευτική ροή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν μπορώ παρά να σκέφτομαι τι επιπτώσεις θα έχει αυτή ε, η αλλαγή για τις γυναίκες και για τους νέους. Δεν θα μιλήσω με στατιστικά στοιχεία, αλλά σαν επιχείρηση δημοσιεύουμε τα δικά μας στατιστικά στοιχεία τον Νοέμβριο του 2014 και βλέπουμε ότι το 85% των τεχνικών θέσεων της εταιρείας πληρούνται από άνδρες και στις γυναίκες διευθυντικές θέσεις δεν ξεπερνάμε το 19%. Θα κάνω ένα πλαίσιο για τη συζήτηση λοιπόν και αν θυμηθείτε κάτι από αυτά τα οποία θα πω σήμερα είναι αυτά τα τρία. Καταρχάς, η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες και φυσικά και οι άνδρες πρέπει να είναι τμήμα της λύσης. Θα ακούσετε αρκετά τα οποία αναφέρθηκαν ίσως και από τις δύο προλαλήσεις. Όπως είχε πει η Μάρια Εντελμέντ, αν δεν σου αρέσει ο κόσμος όπως είναι, μπορείς να τον αλλάξεις. Έχει το καθήκον και την υποχρέωση να το αλλάξεις. συνεργαζόμενοι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε ε, τα προβλήματα αυτά και θα καταστήσουμε τη θέση μας πιο ισχυρή. Εμείς ε, έχουμε δανειστεί τη υγεία από τα παιδιά μας ε, και καλό θα είναι να μάθουμε τα παιδιά αυτά να είναι ικανά να δουν ποια είναι η πραγματικότητα. Έχουν υπάρξει αλλαγές και θα υπάρξουν αλλαγές που ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας μας. Το δικό μου όραμα λοιπόν είναι πραγματικά μια υπερκριτική ε, υψηλού επίπεδου οικονομία. Μια τέτοια οικονομία η οποία να συμπεριλαμβάνει τις ανθρώπινες αξίες και αυτό είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει καινοτομία, θέσεις απασχόλησης, περισσότερη καινοτομία, περισσότερες ιδέες. Η τεχνολογία για μας είναι ο στόχος απαιτείται να εκπαιδευθούν περισσότερες γυναίκες έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά ηγετών γυναικών. Ε, επιμένω λοιπόν σε αυτήν την υπερκριτική ε, οικονομία και αντίληψη, μια πλατφόρμα στην οποία η φαντασία θα ξεπερνά τις διαφορετικές πολιτιστικές αξίες και να σας μιλήσω το τι θα μπορούσε να είναι μια τέτοια φτηνή πλατφόρμα. Να δούμε την τεχνολογία σαν κάτι τις γυναίκες να ενισχύσουν τη θέση τους στην ψηφιακή κοινωνία. Η ελεύθερης χρήση πηγή σαν παράδειγμα. Είναι μια τεχνολογία η οποία θα βοηθήσει. Μπορεί να υπάρχουν ειδικέ εφαρμογές για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου από τις γυναίκες και αυτές ε, οι ανοιχτής πηγής, οι ελεύθερης πηγής, ε, στη, ή μάλλον πληροφορίες και αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μας σήμερα. Το λεγόμενο GitHub θα είναι τα θεμέλια για αυτή την πλατφόρμα, η οποία θα είναι όπως είπα open source ελεύθερης ε, χρήσης της πηγής οι γυναίκες από όλο τον κόσμο θα συνεργάζονται και θα βοηθούν η μία την άλλη για καλύτερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω smartphone και tablets. Υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες θέλουν να, να ταράξουν λίγο τα, τα επίπεδα στα οποία λειτουργούν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες. Εταιρείες όπως η XPRIZE είναι καταλήτες μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν παράδειγμα κάποιος, ε, κάποιες ταμπλέτες σε κάποια απομεμακρυσμένα χωριά και αυτό δεν είναι κάτι μόνο που ε, θα γνωρίζουν τα παιδιά μόνα τους αλλά θα μαθαίνουν ο ένας τον άλλο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ε, του τι μπορεί να γίνει με μια πλατφόρμα C όπου η τεχνολογία θα βοηθά τις γυναίκες μπορούμε να χρησιμοποιούμε και για τις εμπορικές συναλλαγές. Δεν θα υπάρχουν εκεί παραδοσιακές τραπεζικές καταθέσεις. Η εικόνα την οποία έχω είναι το διαδίκτυο των γυναικών. Ένα διαδίκτυο το οποίο θα είναι αποκλειστικά γυναικείο. Χρειάζονται οι εταιρείε της υψηλής τεχνολογίας τις γυναίκες, είναι οδηγοί οι γυναίκες για τις νέες τεχνολογίες στην, στον τομέα του διαδικτύου και στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και στον τομέα των κοινωνικών δικτυώσεων. Η τεχνολογία συνεχίζει να επηρεάζει τη ζωή μας και οι εργαζόμενοι απαιτούν, απαιτείται να έχουν νέες ικανότητες και οι δυνατότητες εργασίας στην τεχνολογία αυξάνονται τρεις φορές πιο γρήγορα από άλλες καριέρες στην Ευρώπη. Οι ρυθμοί της αλλαγής και της καινοτομίας επιταχύνονται και θα πρέπει να είμαστε ατρόμητοι όλοι σήμερα και να διατρέχουμε κινδύνους, να ξεπερνάμε τα εμπόδια, να χαράζουμε νέους δρόμους. 7,3 δις οι κάτοικοι της γης και προβλέπονται να είναι 8 δις την άνοιξη του 24 και οι γυναίκες είναι το 51% της παγκόσμιας οικονομίας. Κι όμως πολλές φορές τις γυναίκες αυτές τις αγνοούμε σε περιπτώσεις κρίσης. Όταν μιλάμε για την ισότητα των φύλων, για να κρίνουμε το τι κάνουμε στις ψηφιακές κοινωνίες, βλέπουμε ότι την κατηγορία αυτή δεν τη θεωρούμε καταλήτη και αποτυγχάνουμε σε αυτό. Είναι τραγική αυτή η άγνοια. Πολλές φορές οι γυναίκες ε, δεν λαμβάνονται υπόψη και όμως η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδης για τα θέματα αυτά. Μην υποτιμάτε σε καμία περίπτωση τις επιπτώσεις ε, που έχουν τα μέσα ενημέρωσης από πλευράς των γυναικών σαν καταλήτης για την αλλαγή. Αν δεν βλέπεις όμως κάτι δεν μπορείς να το αισθανθεί και θα ήταν εύκολο για μένα να μιλήσω για την τεχνολογία, αλλά εδώ ας, ε, ε, ας μιλήσουμε περισσότερο για θέματα οργάνωσης. Ε, οι οργανωτικές αλλαγές και οι πολιτιστικές αλλαγές είναι κάτι το διαφορετικό. Στη ΣΥΣΚΟ οι άνδρες και οι γυναίκες αναζητούν γυναίκες συμμάχους έτσι ώστε να είμαστε τολμηροί και να ακολουθήσουμε δρόμους που κανείς στην επιχείρηση δεν έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα. Ε, το πρόγραμμά μας Men for Inclusion, ε, άνδρες για την συνεργασία και τη συμπερίληψη των γυναικών. Θα είναι ένα καύσιμο για την καινοτομία και για τις γυναίκες τον καλύτερό τους ρόλο. Θα είναι κάτι το μετρήσιμο. Είναι κάτι το οποίο θα προκαλέσει περισσότερη καινοτομία. Θα χρειαστούμε πέντε χρόνια. Είναι ένα ταξίδι μακρύ αλλά αυτό το οποίο όμως βλέπουμε στο τέλος είναι καλύτερες ευκαιρίες για προσλήψεις, για ανάπτυξη, μεγαλύτερη αλληλοεπίδραση ανδρών γυναικών, επιλογές για τις γυναίκες, καλύτερα αποτελέσματα για την εταιρεία, τη ΣΥΣΚΟ. Και ακριβώς εμείς θέλουμε να κρατήσουμε τα ταλέντα αυτά. Ε, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει απλά να εκπαιδεύουμε σωστά, αλλά να κρατάμε. Όπως είπε η Κάθριν Άσκροφτ, ερευνήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ότι οι γυναίκες που ασχολούνται με τα τεχνικά είναι ισχυρές γυναίκες και οι άνδρες που ασχολούνται με τα τεχνικά δεν είναι ο εχθρός όμως υπάρχουν κοινωνικές προκαταλήψεις οι οποίες μας επηρεάζουν όλοι. Πρέπει να αναλάβουμε δράση λοιπόν από κοινού όλοι μαζί. Έχουμε βιώσει ε, τα προβλήματα που υπονομεύουν την αίσθηση εμπιστοσύνης που έχει η γυναίκα για τον εαυτό της. Γι' αυτό λοιπόν τώρα θα σας βάλω δουλειά. Εννέα συστάσεις. Έχω εννέα συστάσεις, κάποιες από αυτές έχουν ήδη αναφερθεί από σας πέρα από θέματα διαφθρωτικά όπως γονική άδεια, μητρική άδεια, πατρική άδεια, σωστή εκπαίδευση, κατάρτιση κτλ. Καταρχάς, μια εκστρατεία ενημέρωσης που δείχνει άνδρες να προωθούν τις γυναίκες. Δεύτερον, ένα, μπορεί κανείς να παράγει ας πούμε ε, κινηματογραφικά έργα με τίτλους όπως «Αυτή θα τα καταφέρει» Υπάρχει κάτι τέτοιο που δείχνει πόσο έχουν ανέβει οι γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε γυναίκες οι οποίες έχουν ηγετικέ θέσεις ιστορικά στα σχολεία, στα πανεπιστήμια κτλ. Έχουμε πολύ ωραίες τέτοιες ιστορίες, πρέπει να δείξουμε το τι συμβαίνει. Ε, επισκέφτηκα την επιμελήτρια ενός γυναικείου μουσείου στις Ηνωμένε Πολιτείες και αναφέρθηκε σε κάποιες γυναίκες από τον μεγάλο υπολογιστή και όταν χρειάστηκε να αναγνωριστούν οι, άνθρωποι οι οποίοι είχαν εφεύρει τους αλγορίθμους ε, σε επίπεδο ηλεκτρονικού υπολογιστή η απάντηση δυστυχώς ήταν ότι δεν ήταν πραγματικά πρόσωπα αλλά ηλεκτρονικά μοντέλα ενώ αυτό φυσικά ήταν εντελώς λάθος απλά δεν χώραγε στα στοιχεία του υπολογιστή. Τώρα επίσης να υπάρξει ένα βραβείο Νόμπελ για τις γυναίκες να υπάρξει επίσης επιμονή και υπογράμμιση της δυνατότητας ανάληψης ευθυνών για τα πρόσωπα και επαφή στενή ανάμεσα στα διαφορετικά πρόσωπα. Να στηριχθούν επίσης αγώνες για γυναίκες και κορίτσια με άνδρες ως προπονητές. Επίσης να ενθαρρύνουμε την κατάρτιση για απόκτηση ικανοτήτων από τις γυναίκες στη μέση και στο τέλος της σταδιοδρομίας τους. Εμείς το έχουμε πει στα πλαίσια του pipelining, δεν μ' αρέσει βέβαια ο όρος αυτός, αλλά όταν κάποιος είναι 30, 40 ή 50 ετών και θέλει να μάθει πράγματα για την τεχνολογία, έχουμε την αίσθηση ότι τους αγνοούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι λοιπόν ποτέ αργά θα λέγεται η εκστρατεία αυτή. Ας το κάνουμε λοιπόν. Θα πρέπει επίσης να ε, έχουμε στρογγύλες τράπεζες ε, με άνδρες και γυναίκες στις μεγάλες διασκέψεις. Ε, υπάρχει πλειοψηφία ανδρών στην τράπεζα και η πλειοψηφία του κοινού είναι γυναίκες. Και τέλος να ενισχύσουμε τα λεγόμενα pitch, ε, ε, δηλαδή το στήσιμο πριν το shoot, οι γυναίκες να βοηθηθούν στην επιχειρηματικότητά τους. Αυτή τη στιγμή οι γυναίκες λοιπόν μπορούν να δράσουν, εμπλέκονται και ε, τότε σε αυτή την περίπτωση θα ασχοληθούν και αυτό είναι το μέλλον του ίντερνετ από τις γυναίκες για τις γυναίκες. Όταν έχουμε το σωστό ταλέντο θα προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, είναι ευγενής ο στόχος μας να ζητήσουμε από τους άνδρες να γίνουν σύμμαχοι και να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα πλανήτη 50% 50% άνδρες γυναίκες μέσα της πλατφόρμας ΣΥ. Έτσι θα αποκαταστήσουμε και τα κενά στην διπλή παραγωγικότητα και όχι μόνο στην έλλειψη των γυναικών και ιδιαίτερα στον υπόλοιπο κόσμο γυναίκες που πεθαίνουν γιατί δεν έχουν τα σωστά φάρμακα. Λοιπόν πρέπει να τολμήσουμε, η Ευρώπη έχει κάθε δυνατότητα να είναι πρόδρομος σε αυτόν τον κόσμο, ας δράσει τώρα.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 en dicho informe para posteriormente pasar al debate con el resto de ponentes en la sombra de los grupos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομιλήτριες. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακότατα αυτά που μας είπατε και πολύ εξισορροπημένες οι παρουσιάσεις. Μας αναφέρατε πληθώρα παραδειγμάτων όπου βλέπουμε την πλήρη διάσταση της ε, ενδυνάμωσης του ρόλου των γυναικών. Και πρέπει να δούμε και το υπόβαθρο, να δούμε γιατί θέλουμε αυτή την έκθεση, γιατί πρέπει να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε. Η ψηφιοποίηση αυτή τη στιγμή είναι κάτι επαναστατικό, αλλάζει εκ θεμελίων την κοινωνία και φυσικά έχει θετικά και αρνητικά, έχει πολλές ευκαιρίες όμως που πρέπει πρέπει να αδράξουμε. Ιδιαίτερα με την χρήση δημοκρατικής πλατφόρμας, όπως μας ε, είπατε εσείς ε, κυρία Σχάμ, για να δημιουργήσουμε μία ε, οικονομική σφαίρα με περισσότερες εκφάνσεις, με περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αλλάζει η αγορά εργασίας, όπως είπατε και εσείς ε, κυρία Μπεζέ. Επίσης πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι όμως ε, που περιέχονται και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή έχουμε δουλέψει πάρα πολύ ιδιαίτερα για να καταπολεμηθεί η έμφυλη βία και να δούμε τι βήματα μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να καταπολεμήσει αυτό το πρόβλημα που έχει εμφανιστεί, όχι από το διαδίκτυο που έχει ενισχυθεί όμως και επιδεινωθεί από το διαδίκτυο. Μιλώ για τη βία κατά των γυναικών που λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις τώρα στο διαδίκτυο. Είναι πιστεύω σωστός ε, χρόνος να το συζητήσουμε αυτό γιατί βρισκόμαστε στην αφετηρία ε, της ψηφιακής ατζέντα, του ψηφιακού θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χρειάζεται λοιπόν να συζητήσουμε πώς ε, μπορούμε να στηρίξουμε την βιώσιμη ψηφιοποίηση διαφοροποίηση της κοινωνίας μας, όμως δεν έχει συζητηθεί η ισότητα, δεν έχει τεθεί ως ένας από τους βασικούς επιλώνες αυτού του οικοδομήματος. Και βλέπουμε ε, ότι υπάρχει λοιπόν αυτή η έλλειψη. Θέλουμε να συμπεριληφθούν και οι γυναίκες ε, στην ε, ψηφιακή αυτή επανάσταση και πιστεύω πως πρέπει η ισότητα να είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές. Αυτό συνεπάγεται τη συμπερίληψη των γυναικών σε όλους τους τομείς. Θα ήθελα τώρα να ξεχωρίσω ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην έκθεση. Εσείς πιστεύω ότι αναφέρετε πολλά περισσότερα Βέβαια όμως ενδεικτικά θα σας αναφέρω ορισμένα θέματα που θεωρώ σημαντικά σε αυτό το έγγραφο εργασίας. Όταν μιλούμε καταρχάς για δημοκρατία πρέπει να μην ξεχνάμε και την εκπαίδευση, την κατάρνηση και την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επίσης ε, πρέπει να, να ε, διασφαλίζουμε μία βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να δούμε τρόπους προσέγγισης. Ως ε, εισηγήτρια συζητώντας την ε, έκθεση αυτή είδα πάρα πολλά πάρα πολλές πληροφορίες, έλαβα πολλές πληροφορίες από τους συναδέλφους, από εσάς ακόμα περισσότερο. Η ψηφιοποίηση της ε, κοινωνίας είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο ως μια δημοκρατική πλατφόρμα. Μια τέτοια πλατφόρμα δίνει πολύ μεγάλη δύναμη, ιδιαίτερα στις ε, γυναίκες. Δίνει δύναμη σε όλες τις περιθωριοποιημένες ομάδες. Οι γυναίκες αποτελούν το 51% του πληθυσμού της γης και δυστυχώ ε, όμως αυτό το ποσοστό δεν διαφαίνεται. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την ψηφιοποίηση έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών. Ε, όσον αφορά την αγορά εργασίας τώρα, μας είπατε ε, κι εσείς για το ποσοστό συμμετοχής ε, των γυναικών στην, στις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής. Μόνο το 15% των απασχολούμενων σε αυτόν τον τομέα είναι γυναίκες. Και φανταστείτε πόσες πολλές θέσεις απασχόλησης θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και να καλυφθούν από γυναίκες. Είναι μια τεράστια ευκαιρία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε οι γυναίκες να ε, μπουν σε αυτόν τον χώρο. Κάθε χρόνο δημιουργούνται 120.000 νέες θέσεις εργασίας στον τομέα της ε, επικοινωνίας και της πληροφορικής και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Επίσης αναφερθήκατε στην υποεκπροσώπηση των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ιδιαίτερα στον χώρο της πληροφορικής και της επικοινωνίας. Μας είπατε για τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων εταιριών. Όντως υπάρχει πρόβλημα εκεί, υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να συζητηθεί το πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στις γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτόν τον χρόνο. Και Μονίκα μας έδωσε πάρα πολύ ε, εύστοχα παραδείγματα για το πώς μπορούν οι γυναίκες να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια. Η ψηφιοποίηση θα επηρεάσει όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, θα δημιουργήσει τις θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό θέμα αυτό, ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Επίσης, η κυρία Μπεζό μας αναφέρει το παράδειγμα του Uber, και αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για τις συνθήκες εργασίας και για το πόσο μπορούμε να διασφαλίσουμε σωστές συνθήκες εργασίας ε, στην ψηφιακή αγορά. Υπάρχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια στρατηγική που θα εξισορροπήσει καλύτερα την επαγγελματική και προσωπική ζωή. Εκεί έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε την αισθητική αυτή για να δώσουμε καλύτερη πρόσβαση στην αγορά στις γυναίκες και πρέπει αυτό να το ε, διαμορφώσουμε. Επίσης άκουσα πως αναφέρατε τη σημασία της εκπαίδευσης. Δεν ε, είναι σημαντικό μόνο να μπουν οι γυναίκες στην ε, συζήτηση, πρέπει να συμπεριληφθούν τα ψηφιακά θέματα στον γενικότερο κύκλο εκπαίδευσης στα σχολεία, για παράδειγμα, στα πανεπιστήμια, χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση για ψηφιακά ζητήματα, διότι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα επηρεάσει όλους μας αυτή η αλλαγή. Επίσης, η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη είναι προφανές πως χρειάζεται ε, πολυμορφία. Πρέπει να δώσουμε πολλές διαστάσεις στην οικονομία μας έτσι ώστε αυτή να γίνει βιώσιμη. Και εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις γυναίκες που υποεκπροσωπούνται γιατί αυτές θα αλλάξουν την κοινωνία μας. Έχουν το δυναμικό να το κάνουν τα επόμενα χρόνια. Χρειάζεται όμως επίσης να δούμε και τις δυνατότητες χρηματοδότησης για τις νεοσύστατες εταιρείε. Ε, έχουμε το επενδυτικό σχέδιο Juncker για το πώς θα κατανεμηθούν αυτοί οι πόροι και χρειάζεται επίσης να κατανεμηθούν και με βάση κάποια κριτήρια και πρέπει εκεί να ληφθεί υπόψη η υποεκπροσώπηση των γυναικών. Επίσης χρειάζεται να δούμε τα θετικά παραδείγματα των νέων γυναικών επιχειρηματιών οι οποίες ε, κατάφεραν να πετύχουν σε έναν ανδροκαρτούμενο κόσμο και πρέπει να προωθηθούν αυτά τα παραδείγματα, να προβληθούν έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα και σε άλλες γυναίκες. Τέλος, εδώ θα επανέλθω σε αυτά που ανέφερε η κυρία Σχάμ, είναι το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών. Πρέπει να το συζητήσουμε ανοιχτά, πρέπει να αναφερθεί και στην έκθεση, να δείξουμε ότι υπάρχουν προβλήματα με τον εκφοβισμό, με τη ρητορική μίσους, ε, στο διαδίκτυο, ότι χρησιμοποιείται το διαδίκτυο ως μια πλατφόρμα για να ενισχυθούν τα πατριαρχικά και ανδροκρατούμενα κοινωνικά πρότυπα και χρειάζεται να δημιουργηθούν ε, όργανα που θα προσθεθούν στα ήδη υπάρχοντα στήριξη, για παράδειγμα, στην κοινωνία των πολιτών, καλύτερη κατάρτιση όπως προτείνατε στα, στις αστυνομικές ε, αρχές, καλύτερη κατάρτιση στο χώρο της ε, εκπαίδευσης. Επίσης, όπως είπατε και στην αρχή, πρέπει οι γυναίκες να δείξουν αλληλεγγύη μεταξύ τους, πρέπει να δικτυωθούν έτσι ώστε να ε, μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις εξιστικές επιθέσεις. Ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα δίκτυα νέων και ε, μεγαλύτερων γυναικών. Όπως είπε σε Μονίκ, ποτέ δεν είναι αργά για να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο, για να το χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να προβάλλουμε αντίσταση σε αυτές τις επιθέσεις. Ακούστηκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες λοιπόν και ελπίζω και οι συνάδελφοί μου να μου δώσουν ακόμα περισσότερες έτσι ώστε να ε, διαμορφώσουμε την έκθεση. Γι' αυτό λοιπόν με χαρά μου θα περιμένω τα σχόλιά σας, την συμμετοχή σας και επίσης θα ήθελα να συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών ακόμα περισσότερο. Όλοι οι ε, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα νέα δεδομένα και έτσι ώστε να αλλάξει το ψηφιακό θεματολόγιο και έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος των γυναικών εκεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ρέντνερ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την συζήτηση αν θέλετε με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων η κυρία Λεγκρίπ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω ολόθερμα τις τρεις ομιλήτριες της σημερινής ακρόασης. Ήταν συναρπαστικές, συναρπαστικές τρεις παρουσιάσεις. Και το εννοώ. Κρίμα, κρίμα. Όσοι δεν μπορούσαν να βρουν χρόνο για να έρθουν ε, σήμερα μαζί μας, ε, έχασαν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Βεβαίως επειδή υπάρχει το αρχείο στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου μπορούν να τα ακούσουν στη συνέχεια. Ήσασταν εξαιρετικές και οι τρεις. Χαίρομαι επίσης ε, με όλες αυτές τις ιδέες της εισηγήτριάς μας. Μόλις μας έκανε μια ακριβέστατη παρουσίαση όπου φαίνεται η θέλησή της να τροφοδοτήσει ε, να τροφοδοτήσει και να δώσει μια νέα δυναμική ε, με τις ιδέες της στη συζήτησή μας. Εγώ θα ήθελα να πω πως και τώρα παραπέμπω στον τίτλο της σημερινής ακρόσης ε, χειραφέτηση των γυναικών στην ψηφιακή εποχή. Πρόκειται για μια τρίτη ε, βιομηχανική επανάσταση η ψηφιακή επανάσταση ή επανάσταση χάρη στην οποία τα κορίτσια, 9 γυναίκες θα μπορέσουν να κατακτήσουν το χώρο που δικαιούνται, να διαδραματίσουν το ρόλο που τους αναλογεί στην κοινωνία, να κατακτήσουν την ισότητα με το άλλο φύλλο. Στις προηγούμενες επαναστάσεις οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Υπέστησαν πολλές ζημιές οι γυναίκες και δεν μπορούσαν να μετάσχουν πλήρως στις, σε αυτές τις επαναστάσεις. Αυτή τη φορά όμως δεν πρέπει να χάσουν αυτή την ευκαιρία. Είναι η καταπληκτικότερη ευκαιρία που είχαν ποτέ, όπως μας είπε σωστά η κυρία Μπερζέ, να κατακτήσουν αυτό το νέο χώρο για την πολιτική και οικονομική τους χειραφέτηση. Είδαμε πολύ πρόσφατα στην Αραβική Άνοιξη ότι ε, μια πολιτική ε, χειραφέτηση. Ε, φυσικά ε, μπορούμε να ακούσουμε ε, τα αντίθετα επιχειρήματα, αλλά για πρώτη φορά στην παγκόσμια πολιτική σκηνή πρώτη φορά πήραν την εξουσία κατά αυτόν τον τρόπο στα χέρια τους οι νέες γυναίκες Βλέπουμε επίσης ε, στα χωριά, στα αγροκτήματα, γυναίκες να ε, αλλάζουν το ρόλο τους, να βρίσκουν τρόπους ε, να ε, συμμετάσχουν στον εμπορικό ε, βίο μέσω αυτής της οικονομικής χειραφέτησης σε χώρους όπου δυσκολεύονταν αιώνες οι γυναίκες να βρουν τη θέση που μπορούν να διεκδικήσουν πλέον έχουν νέες ευκαιρίες και εσείς και η συγγήτριά μας ε, σωστά ε, δίνετε τη μεγαλύτερη έμφαση στην παιδεία, στην εκπαίδευση. Υπάρχει βέβαια και η διάσταση της ε, αυτοπεποίθησης. Έχει ιδιαίτερα μεγάλο ειδικό βάρος για τη γενιά, μου ούτως ή άλλως, αλλά και για τις, τα κορίτσια και τις γυναίκες. Έχω τρία παιδιά, τρία κορίτσια ε, μάλλον, συγγνώμη, ένα αγόρι και δύο κορίτσια και βλέπω ότι υπάρχουν διαφορές, δηλαδή με άλλο τρόπο συμμετέχουν οι κόρες μου ε, στον ψηφιακό χώρο, δηλαδή αυτή η σεξιστική διάσταση υπάρχει ακόμη και νομίζω ότι αυτό φαίνεται και από μελέτες. Έχουν μια πιο κοινωνική προσέγγιση οι γυναίκες, ε, κοινωνικά φόρ, ε, ανταλλαγές απόψεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό προτιμούν ε, τα κορίτσια. Καλά και είναι οι τρόποι κατανάλωσης φυσικά με την ψηφιακή εποχή. Αυτό ικανοποιεί ιδιαίτερα τις νέες γενιές των ε, κοριτσιών και νέων γυναικών, όμως πέραν αυτού θα έπρεπε να κατακτήσουν και χώρους εξουσίας στις επιχειρήσεις, παραδείγματος χάρη, να μπορέσουν να ασκήσουν επιρροή, να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση αυτού του νέου κόσμου, να μην ε, έχουμε παθητική προσέγγιση, όχι με ενεργητικό τρόπο να δραστηριοποιηθούμε, να βάλουμε και εμείς το λιθαράκι μας να συμμετάσχουμε και όχι μόνο να δεχόμαστε τις νέες εξελίξεις και να τις ακολουθούμε, αλλά να τις διαμορφώνουμε. Ε, αυτό θα το επιτύχουμε με την επιμόρφωση με την κατάρτιση για τα, τους νέους τρόπους επικοινωνίας για τα νέα ε, κοινωνικά δίκτυα, ούτως ώστε να προβληθεί αυτός ο στόχος ε, για τις γυναίκες, για τα κορίτσια. Και στο παρελθόν βλέπουμε τι γινόταν στον επιστημονικό τομέα και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ε, δεν βρίσκουμε στον επιστημονικό κλάδο και γυναικείες μορφές ε, που ε, πάτησαν σε παρθέν εδάφη και ε, βοήθησαν να ε, επιτευχθούν ε, καταλυτικές αλλαγές στον επιστημονικό τομέα. Αυτό θα βοηθούσε να ανέβει και η αυτοπεποίθηση των γυναικών και να καταπολεμηθεί αυτό το σύνδρομο του φτωχού συγγενή ή εν πάση περιπτώσει το σύνδρομο κατωτερότητας από το οποίο υποφέρουν. Ελπίζω όλες αυτές τις καταπληκτικές ιδέες να τις συμπεριλάβουμε στην έκθεση και στις τροπολογίες μας. Σας ευχαριστώ κλείνοντας και πάλι για τις ε, πολύ καλές ιδέες που μας δώσατε. Ευχαριστούμε κυρία Λεγκρύπ. Η σκιώδης, η συγγήτρια από σοσιαλιστές είμαι εγώ υποφαινόμενη. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω λίγα λεπτά για να επαναλάβω τις ευχαριστίες μου στις τρεις συναδέλφους που πήραν μέρος στην ακρόαση. Να ευχαριστήσω επίσης και για την παρουσίαση της ηγήτριας η οποία αντιμετωπίζει με σφαιρικό τρόπο όλα τα θέματα τα οποία μας ανησυχούν στην παρούσα στιγμή. Το θέμα της ενίσχυσης του ρόλου των γυναικών στον ψηφιακό κόσμο περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά θέματα. Το πρώτο είναι η δυνατότητα που έχουν οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε ό,τι έχει σχέση με αυτό το θέμα και το άλλο είναι η δυνατότητα η οποία υπάρχει να ενσωματώσουμε σε αυτή την προσπάθεια συγκεκριμένες δράσεις. Νομίζω λοιπόν ότι στον τομέα της πρόσβασης είναι σαφές ότι θα πρέπει να αναφέρουμε ότι στα πλαίσια του στρατηγικού προγράμματος για την ισότητα που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2015 να υπάρξει συγκεκριμένη αναφορά σε όλα αυτά όπως η στήριξη στις ε, οργανώσεις των εργοδοτών αλλά και των εργαζομένων που ασχολούνται με θέματα φύλου. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να δούμε ακριβώς τι γίνεται με τα διαφορετικά ταμεία και σε ποιο βαθμό μπορούν να βοηθήσουν την πρόσβαση των γυναικών ή μάλλον να βοηθήσουμε καλύτερα τις γυναίκες οι οποίες ζουν σε γεωργικές περιοχές, σε περιοχές της υπαίθρου. Υπάρχει αναφορά λοιπόν σε όλα αυτά έτσι ώστε τα προγράμματα τα οποία προωθούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία να λαμβάνουν υπόψη τη συγκεκριμένη αυτή κατάσταση για τις γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο σε σχέση με τις γυναίκες που ζουν σε αστικές περιοχές. Κατά τα άλλα δεν έχω να πω παρά συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε η κυρία Λεγκρίπ και η συγκήτρια θα δώσω το λόγο στην ε, σκιώδη συγγήτρια της ομάδας των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλες τις ομιλήτριες για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ακούσαμε. Ήμουν στη Γενέβη λίγο νωρίτερα με μέλη αυτής της Επιτροπής στο συνέδριο και μου έκανε εντύπωση αυτό που είπατε για την εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών, διότι οι περισσότεροι στο πάνελ ήταν άντρες και μάλιστα έγραφαν στα κοινωνικά μέσα για αυτά που κάναμε. Ένα από αυτά που βρήκα πολύ ενδιαφέρον ήταν το, η περίπτωση του Μπαγκλαντές. Ψηφιοποίησαν όλα τα κυβερνητικά τους ε, προγράμματα. Οποιαδήποτε επαφή που θέλει κάποιος να έχει με την κυβέρνηση στο Μπαγκλαντές γίνεται ψηφιακά. Επένδυσαν λοιπόν στις ψηφιακές υποδομές και απόρρια αυτού είναι ότι σε κάποια απομονωμένα χωριά έδωσαν ένα φωτοβολταϊκό πάνελ και ένα τάμπλετ και έτσι ο καθένας από αυτό το χωριό θα μπορούσε να κάνει τις δουλειές του ηλεκτρονικά, να κάνει συναλλαγές στον τραπεζικό του λογαριασμό. Τα πάντα ηλεκτρονικά, μέσω αυτού του τάμπλετ λοιπόν. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτή η ψηφιακή επανάσταση, η ψηφιοποίηση έχει φέρει πολλά θετικά. Ε, ωστόσο είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με τα δεδομένα μας και πώς αυτά χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο. Σίγουρα υπάρχουν καλές περιπτώσεις και κακές περιπτώσεις. Εξαρτάται από τον τομέα. Κάποιοι από εμά βέβαια δεν ασχολούνται τόσο με το διαδίκτυο όσο κάποιοι άλλοι και δεν ενδιαφέρονται για το τι συμβαίνει εκεί τόσο όσο άλλοι. Ε, μπορώ να παρομοιάσω πάντως αυτήν την κατάσταση που επικρατεί τώρα με τη θέση των γυναικών ε, κάποια χρόνια πριν. Τη δεκαετία του 50 οι γυναίκες ήταν στην κουζίνα. Τώρα ε, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Σκεφτείτε λοιπόν τι θεωρούταν κοινωνικά αποδεκτό τη δεκαετία του 50 ή του 60 και πού βρισκόμαστε τώρα. Έχουν λοιπόν αλλάξει πάρα πολλά και τα θέματα αυτά που άλλοτε θεωρούνταν ταμπού έχουν βρει δημόσιο βήμα. Είναι λοιπόν πολύ καλό που επιτέλους μπορούν οι γυναίκες να συζητήσουν δημόσια στο διαδίκτυο θέματα παρενόχλησης, θέματα κακοποίησης, εξιστικής βίας. Και είναι καλό που υπάρχουν αυτές οι φωνές. Και όπου ε, αναφερθήκατε στην ε, φραστική βία που εξαπολύεται εναντίον των γυναικών στο διαδίκτυο. Και εγώ ίδια έχω δεχθεί τέτοια βία στο Twitter, στο Facebook. Το κάνω, ε, όμως συνεχίζω, δεν επηρεάζομαι. Εξωτερικεύω αυτές, ε, αυτή την επίθεση και δεν κλείνομαι στο καβούκι μου. Και πιστεύω εδώ ότι η εκπαίδευση έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Πρέπει να διδαχθούν τα παιδιά στα σχολεία, όχι γράμματα και αριθμούς, να διδαχθούν τις αιτίε πίσω από αυτούς τους αριθμούς, πίσω από αυτά τα στατιστικά στοιχεία, να διδαχθούν το ότι πρέπει να αμφισβητούν, πρέπει να κάνουν ερωτήσεις για να βρουν απαντήσεις. Η παιδεία λοιπόν πιστεύω πως επιδέχεται βελτίωσης και σίγουρα δεν πρέπει να παραμεληθεί. Επίσης, οι ιδιοκτήτες αυτών των ψηφιακών ε, πλατφόρμων, του Twitter, του Facebook, δεν πρέπει να μείνουν αμέτωχοι. Έχουν ηθικό καθήκον να επιτηρούν και να αναφέρουν τέτοια περιστατικά επιθέσεων στις γυναίκες. Πώς μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε ε, τις γυναίκες έτσι ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Η επιχειρηματικότητα είναι ένας προβληματικός τομέας. Υπάρχει ακόμα τεράστιο κενό, υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες. Και αναρωτιέμαι γιατί αυτός ο τομέας δεν είναι ένας τομέας που ενδιαφέρει τις ε, γυναίκες. Ίσως είναι θέμα βιολογίας, διαφέρουμε από τους άντρες, έχουμε διαφορετική προσέγγιση από τους άντρες σε πολλά ε, θέματα. Οι γυναίκες συνεργάζονται πιο εύκολα με άλλες ε, γυναίκες, με ανθρώπους, ενώ οι άντρες είναι περισσότερο ε, μοναχικοί στη δουλειά τους. Υπάρχει λοιπόν μια επιθυμία των γυναικών για συνεργασία και ίσως αυτό θα μπορούσαμε να το ενισχύσουμε. Και ίσως οι εταιρείες θα έπρεπε να βελτιώσουν το εργασιακό τους περιβάλλον. Να σας αναφέρω ενδεικτικά ότι με την Επιτροπή Μεταφορών πήγαμε στο Δουβλίνο στα γραφεία της Google και είδα τα γραφεία τους, ε, υπήρχε άπλετος χώρος, συνεδριάσεων, υπήρχε χώρος όπου μπορούσαν να συζητήσουν οι υπάλληλοι, ήταν όλα ε, πολύχρωμα. Ήταν λοιπόν ένα πολύ όμορφο εργασιακό περιβάλλον και πρέπει να το πάρουμε ως καλό παράδειγμα. Εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε νομοθετήσει και ορισμένα από αυτά τα νομοθετήματα ήταν αποφασιστική σημασία για τι γυναίκε. Η νομοθεσία σχετικά με τον φόρο προστιθέμενη αξία, για παράδειγμα, είναι μια τέτοια περίπτωση όπου νομοθετήσαμε ότι ο ΦΠΑ πρέπει να πληρώνεται τη στιγμή που παράγεται Και υπάρχουν πολλές ε, γυναίκες, μικροεπιχειρηματίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο διαδικτυακό εμπόριο και έχουν μικρές επιχειρήσεις. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα από την νομοθεσία σχετικά με το φόρο προστιθέμενης αξίας σε όλες τις χώρες της Ένωσης. Και προσπαθούν αυτές οι γυναίκες λοιπόν να συνδυάσουν την ε, προσωπική του ζωή με την ε, επαγγελματική τους ε, ζωή, να τρέξουν δηλαδή μία μικρή διαδικτυακή επιχείρηση. Αυτή η νομοθεσία λοιπόν έχει επηρεάσει αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πολύ συχνά είναι στελεχωμένες από γυναίκες. Επίση, μα είπε, ε, Μόνικα, ότι αν δεν ε, μα αρέσει ο κόσμο, πρέπει να τον αλλάξουμε. Και συμφωνώ. Ο πατέρα μου, μάλιστα, μου έλεγε ότι αν δεν σε αρέσει κάτι, ε, ανέλαβε δράση. Κάνε κάτι. Εσύ. Και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που επηρεάζουν τις γυναίκες και όντως χρειάζεται δράση. Μας αναφέρατε τα στατιστικά στοιχεία και τα νούμερα από τη ΣΥΣΚΟ που θεωρώ πως είναι μια πάρα πολύ προοδευτική εταιρεία. Όμως ε, πρέπει να σας πω ότι δεν πιστεύω πως ε, το σύστημα είναι ο εχθρός μας. Πιστεύω πως το σύστημα πρέπει να αλλάξει και δεν νομίζω πως ε, κάποιος ενοχλείται αν έχει μια γυναίκα προϊστάμενη. Πρέπει να κοιτάξουμε πως θα βελτιωθούν οι εργασιακές σχέσεις ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών και πώς θα βελτιωθεί το εργασιακό περιβάλλον έτσι ώστε να γίνει πιο φιλικό προς τις γυναίκες. Και φυσικά συμφωνώ με όσα υπόθηκαν πιο πριν, δηλαδή για την παρενόχληση των γυναικών και για το ότι χρειάζεται ε, δράση. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, όμως ε, πρέπει να προσέξουμε αυτές οι ευκαιρίες να μην χρησιμοποιηθούν εναντίον μας και μας πάνε 50 χρόνια πίσω. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλες που ήρθατε σήμερα εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βέρνερ. Η κυρία Μόρβαϊ. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω ουγγρικά. Μίλησαν ε, οι συνάδελφοι 8-10 λεπτά η κάθε μία. Χθες 2 λεπτά μίλησα και μου επιτέθηκαν όλοι. Ελπίζω να μην ε, ε υποστώ διακριτική μεταχείριση και σήμερα. Λοιπόν, για να περάσω τώρα στην ουσία. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη μητρότητα και το ίντερνετ. Πώς έχει εξελιχθεί αυτή η σχέση και τι εννοώ και γιατί σας τα λέω αυτά. Μία φορά αναφέρθηκε η μητρότητα από την ε, πρώτη ομιλήτρια. Είναι κάτι εξαιρετικό φυσικά το να έχουμε όλη πρόσβαση ε, στο διαδίκτυο. Μπορούμε να κάνουμε chat Και όσες δεν θέλουν να είναι μητέρες ή το έχουν μετανιώσει μπορούν να μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα και να λένε τον πόνο τους. Εγώ είμαι νομομαθής και ειδικεύομαι στα ζητήματα κακοποίηση των παιδιών. Μπορώ να σας πω Λοιπόν, το ότι όταν κάποιος το έχει μετανιώσει που έκανε παιδί, και ε, εκφράζει αυτό που νιώθει στο ίντερνετ, αυτό είναι και αυτό κακοποίηση του παιδιού. Μια μάνα η οποία το λέει στο διαδίκτυο ότι έχει μετανιώσει που έκανε παιδί και το λέει στις άλλες που επίσης ε, νιώθουν το ίδιο, θα έπρεπε να καταγγέλλεται. Εγώ εδώ και 25 χρόνια, ε, μάλλον έκανα παιδιά πριν από 25 χρόνια και ποτέ δεν το μετάνιωσα. Εντάξει, υπάρχουν και δύσκολες στιγμές στη μητρότητα και νιώθει κάποιος ε, απομονωμένος στο ρόλο της μητέρας, του γονιού. Και μπορεί όντω αυτό να είναι πάρα πολύ δύσκολο, κυρίως για τις μητέρες μικρών παιδιών. Και φυσικά μπορεί να σας βοηθήσει το ίντερνετ για να νιώσετε λιγότερο απομονωμένες. ή για να συνεχίσετε να εργάζεστε, γιατί μπορεί κάποιος να εργαστεί στο διαδίκτυο, το ίδιο ισχύει και για τους ε, άντρες, μπορούν να είναι σε επαφή με το, την εταιρεία τους. Φυσικά το ίντερνετ μπορεί να βοηθήσει τις γυναίκες για να μπουν ε, στην αγορά εργασίας. για να μην νιώθουν τόσο απομονωμένες όταν κάνουν παιδί. Μπορεί να είναι θετικό το διαδίκτυο για την κοινωνική ζωή κάποιου, όμως προσοχή μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Όταν συναντιόμαστε με τους ε, φίλους ε, στην πραγματικότητα, όχι ε, εικονικά, είναι πολύ καλύτερα, έτσι δεν είναι. Ή μπορεί κάποιος να πάει να επισκεφτεί ένα μουσείο επιγραμμικά. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ε, μπορεί μια μητέρα με το μικρό της το παιδί να δυσκολεύεται να πάει στο μουσείο. Όμως μπορεί στο ίντερνετ να επισκέπτεται εικονικά το ένα μουσείο. Βοηθάει το ίντερνετ, δεν λέω. Όταν περνάει η κρίση όμως, ε, μητρώντας μια γυναίκα, πρέπει να τη βοηθήσουμε αυτή τη γυναίκα και εκείνη και το παιδί. Αλλά δεν γίνεται να το μετανιώνει κάποιος. Αν το νιώθει κάποιος πρέπει να ζητάει βοήθεια. Πρόκειται για κακοποίηση του παιδιού και πρέπει να, να μας βοηθήσουν οι επαγγελματίες. Και φτάνω τώρα στην ερώτησή μου που απευθύνω και στις τρεις σας. Μπορεί το ίντερνετ να βοηθήσει αυτές τις γυναίκες. Πώς μπορούμε να τις διαπαιδαγωγήσουμε αυτές τις γυναίκες στην Ουγγαρία. Υπάρχουν δίκτυα γυναικών που βοηθούν άλλες γυναίκες όταν έχουν προβλήματα. Α, έχω και μια άλλη ερώτηση για τις ηλικιωμένε γυναίκες. Δεν απειλούνται από την απομόνωση και εκείνες. Όταν εκείνες ήταν στο σχολείο δεν υπήρχαν όλα αυτά, ούτε υπολογιστές, ούτε το ίντερνετ. Πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε ούτως ώστε να υποφεληθούν και εκείνες τώρα για να μην νιώθουν τόσο μόνες και απομονωμένες. Μπορεί κάποιος σε μια προχωρημένη ηλικία να φτιάξει μια εταιρεία. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Γιάλα θέλει να παρέμβει, αλλά δύο λεπτά. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Για να απαντήσουν και οι τρεις ομιλήτριες. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα αυτό, γι' αυτό πέρασα η σχέση της γυναίκας με την ψηφιακή γενικά οικονομία. Θα ήθελα να ρωτήσω δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, με ποιον τρόπο Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αυτές οι ψηφιακές πλατφόρμες, ιδιαίτερα στη λεγόμενη συνεργατική οικονομία. Ε, και πώς κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει τις συνθήκες εργασίας και πώς μπορεί να επηρεάσει επίσης ε, την ενσωμάτωση των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία και θα ήθελα να μάθω επίσης και τι δυνατότητες μπορεί να έχουμε για να υπάρξει μια ρήτρα εγκάρσια θα έλεγα για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της ε, εφαρμογής μέτρων στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας για τις γυναίκες, δηλαδή περιεχόμενο ψηφιακό, ε, η βία εις βάρος των γυναικών και η προστασία των προσωπικών δεδομένων και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν οι γυναίκες και ακόμα και οι μεγάλες ηλικίε ε, πώς θα μπορέσουν να μάθουν ακριβώς και να ενσωματωθούν στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας. Είναι αλήθεια ότι το να μάθουν οι γυναίκες να εργάζονται στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας είναι ο στόχος. Ευχαριστώ κυρία Γιάλα. Έχουμε 8 λεπτά στη διάθεσή μας μόνο και γι' αυτό θα ήθελα με πάρα πολύ συνθετικό τρόπο Ξέρετε έχουμε μάθει εμείς ε, στην Ολομέλεια να μιλάμε για το θέμα της κατάστασης της Ευρώπης για ένα λεπτό και να λέμε αυτό που θέλουμε να πούμε. Λοιπόν δεν είναι οι ίδιες συνθήκες αλλά θα ήθελα να είχαμε πολύ περισσότερο χρόνο αλλά θα πρέπει να τελειώσουμε στις 12.30 εφόσον εσείς θέλετε να στείλετε κάποιες σκέψεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις οι οποίες έγιναν πριν γραπτά, είμαστε στη διάθεσή μας να τις μοιράσουμε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Θα δώσω το λόγο, θα ξεκινήσω με την κυρία Σραμ. Θα απαντήσω στη μητρική μου γλώσσα, διότι έτσι είμαι πιο άνετη. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας. Είναι πραγματικά πολύ σαφές το τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε οι γυναίκες να στηριχθούν σε αυτή την ε, ψηφιακή κοινωνία, να στηριχθούν και να ενισχυθεί ο ρόλος τους. Μας ε, ρωτήσατε πόσο μπορούν ε, να ενεργήσουν οι πιο ηλικιωμένες γυναίκες έτσι ώστε να προσαρμοστούν. Σίγουρα Επίσης, ε, τι γίνεται στην ε, περίπτωση που οι γυναίκες μετανιώνουν ε, για το γεγονός ότι έκαναν παιδιά. Θεωρώ πως είναι απόλυτα θεμητό και είναι δικαίωμα των γυναικών να μπορούν να πούν κάτι τέτοιο. Εντάξει, το, τα παιδιά θα το καταλάβουν ή όχι, όμως πιστεύω πως είναι αναπόσπαστο κομμάτι του δημόσιου διαλόγου και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ορισμένες γυναίκες επέλεξαν αυτόν τον ίσως ακραίο τρόπο να εκφραστούν. Εντάξει, πολλούς ενοχλεί αυτό το πράγμα, όμως είναι ένα από τα θέματα τα οποία οι γυναίκες δεν τολμούσαν να συζητήσουν πριν από μερικές δεκαετίες και έχει δημιουργηθεί ένας χώρος πλέον ώστε να μπορούν να το πράξουν αυτό. Η μελέτη αυτή, εντάξει, προέρχεται από το Ισραήλ, οπότε ίσως γι' αυτό έχετε πρόβλημα, αλλά σίγουρα κάθε μητέρα έχει το δικαίωμα να εκφραστεί όπως εκείνη επιθυμεί και έχει το δικαίωμα να μην είναι μόνη της και απομονωμένη σε αυτές τις σκέψεις της. Και αυτό έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν τα κοινωνικά μέσα και αυτό πρέπει εμείς ως κοινωνία να στηρίξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπερζέ. Λοιπόν, πολύ γρήγορα για να απαντήσω στο πρώτο ερώτημα για τη σχέση ανάμεσα στη μητρότητα και το διαδίκτυο. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για την, γενικά για τους γονιούς, ε, γονείς και όχι για τις ε, μητέρες, ε, διότι αφορά και τους άντρες, δηλαδή ποια υποστήριξη μπορεί να προσφέρει το διαδίκτυο στους γονείς Μιλήσατε για την Αραβική Άνοιξη. Τι έγινε, παρατηρήθηκε ότι το ίντερνετ γινόταν ένα, ένα ζωντανός, φανταστικός χώρος ε, θεοποιήθηκε, γκομιάστηκε το διαδίκτυο τότε ως ε, δημοκρατικός θεσμός. Ε, όταν βλέπουμε τώρα το λόγο, ε, τη ρητορική μίσους, ε, αυτό δεν αλλάζει τίποτα στη φύση του εργαλείου. Παραμένει ένα δημοκρατικό εργαλείο, όμως θα πρέπει να το ελέγξουμε ως προς το περιεχόμενο που, που δημοσιεύεται. Αν εκφράσετε μια γυναίκα σε ένα κοινωνικό φόρουμ, ποιο πρόβλημα υπάρχει. Το αντίθετο είναι πολύ καλό διότι καταπολεμά την απομόνωση που νιώθει ε, κατά τη διάρκεια της κοίησης ή μετά και εκεί μπορούν να τους βοηθήσουν άντρες και γυναίκες να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα όταν υπάρχει αυτή η ρήξη όπως το είπατε. Τώρα, ε, όπως και για τις μητέρες έτσι και για τις ε, ηλικιωμένες γυναίκες υπάρχει αυτή η ανάγκη επί εκπαίδευσης από, την, από μικρή ηλικία αλλά και επιμόρφωσης ηλικιωμένων ανθρώπων ε, και ούτως ή άλλως αυτό είναι κάτι που γίνεται ήδη. όλα ένα και περισσότερο. Για την συνεργατική, την κοινωνική οικονομία θα έλεγα στην αρχή πως ανανεώνεται η σχέση που έχουμε με την εργασία μέσα από το διαδίκτυο. Ε, δεν θα είναι απαραίτητα μισθωτή πλέον η εργασία μας, ε, θα σχετίζεται περισσότερο με την επιχειρηματικότητα. Έτσι θα έχει πρόσβαση μεγαλύτερη ε, στη δουλειά η γυναίκα. Αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο σε σχέση με το καθεστώς του μισθωτού ή όχι. Ζητώ συγγνώμη που τα λέω τόσο γρήγορα, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Για την ιδιωτική ζωή, αντίθετα, είπε ο ότι είναι η ιδιωτική ζωή μια παρένθεση της ιστορίας και τελικά η ιδιωτική ζωή δεν χρειάζεται, δεν χρήζει προστασίας σήμερα. Το αντίθετο πιστεύουν πολλοί φορείς ε, του κοινωνικού βίου, είναι η ιδιωτική ζωή μια κατάκτησή μας, ένα επίτευμά μας και δουλειά μας είναι να ε, διαφυλάξουμε αυτό το επίτευγμα. Σε επιφυλακή πρέπει να είμαστε γρήγοροι γιατί μπορεί να εκτεθεί, να ε, ε, τεθεί να γίνει ε, αντικείμενο εμπορίου ιδιωτική μας ζωή εάν δεν προσέξουμε. Ξαναλέω ότι ε, απαραίτητη είναι η πρόσβαση στη σωστή πληροφόρηση η προστασία των ατομικών δεδομένων, η προστασία της ιδιωτικής ζωής ε, δεν είναι κάτι που αντιβαίνει στο ίντερνετ. Το αντίθετο συμβαίνει. Για να κλείσουμε τώρα θα ακούσουμε την κυρία Μόρβαη. να μου λέω εγώ προς την κυρία Μόρβαη. Θέλω να σχολιάσω μόνο τελευταίο ερώτημα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ίντερνετ για να κάνουμε κάτι θετικό για τους γονείς και για τους ηλικιωμένους. Βεβαίως, ε, καταφατικά θα σας απαντήσω. Όταν ήμουν στο Μπουτάν, ε, το είδα. Ε, ε, κοινοτικά κέντρα μπορείτε να ιδρύσετε όπου τα παιδιά, οι γυναίκες μπορούν να κάνουν ε, μαθήματα. Το ίδιο ισχύει και για τους ηλικιωμένους να κάνουν συνεδρίες ενημερωτικές ούτως ώστε να προωθήσουμε την κατάρτιση στο ιστορικό μιας κοινότητας. Αυτό και μπορεί και θα έπρεπε να υπάρχει κυρίως ε, για την Ήπεθρο. Αυτό που, μας, ε, συζητούσαμε νωρίτερα. Μεγάλη, καταπληκτική ευκαιρία. Άλλο παράδειγμα. Μία εργαζόμενη γυναίκα που έχει παιδιά μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευελιξία και να δουλεύει από το σπίτι. Εμείς το κάνουμε στη δική μας εταιρεία δεν είσαστε υποχρεωμένοι να έρθετε να, στο γραφείο για να ε, δουλέψετε. Στην IBM ε, ε, έχουμε και ένα φιλμ για την εργαζόμενη μητέρα. Ξυπνάνε, πάει ο άντρας στη δουλειά, αυτή κάθεται πάνω και συνεχίζει να δουλεύει. Είναι πιο ευέλικτη η διαχείριση του χρόνου. Αυτή είναι πολιτική της εταιρείας. Το τελευταίο που ήθελα να πω του διαρθρωτικού χαρακτήρα θέλετε να μιλάμε και για τη μητρότητα και για την πατρότητα και όλοι να συμμετάσχουν στην ε, λύση του προβλήματος ε, και στις δράσεις που αναλαμβάνονται. Δηλαδή και η γυναίκα και η μητέρα και ο πατέρας να το κάνουν και να μην ε, νιώθουν ότι πρέπει να καλύψουν το κενό αυτής της απουσίας τους, να έχουν την προαγωγή που τους αξίζει και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Κοινοτικά κέντρα, ναι, ναι, εκπαίδευση κατάρτιση, επιμόρφωση στο ίντερνετ, ναι, ναι, να σας βοηθούν άλλοι στο διαδίκτυο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και πολλά εκπαιδευτικά επιγραμμικά κέντρα για αυτούς τους σκοπούς. Σας ευχαριστώ για να κλείσει η συζήτηση η συγγήτρια για δύο λεπτά. Δεν χρειάζομαι δύο λεπτά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και τις τρεις εξαιρετικές ομιλήτριες. Είναι η αρχή στις 22 Οκτωβρίου. Θα έχουμε ένα δείπνο εργασίας μετά τη συνεδρίαση. Θα σας στείλουμε μία πρόσκληση έτσι ώστε να μπορέσουμε όλα αυτά ε, να τα εξετάσουμε και ελπίζω η συζήτηση να ήταν ενδιαφέρουσα για όλους. Λοιπόν, διακόπτουμε εδώ, θα συνεχίσουμε στις 3.